Καλύτερε προετοιμασία για την προστασία των ε, συμπολιτών μα για τι μελλοντικέ υγειονομικέ απειλέ. Σα ευχαριστούμε κυρία Επίτροπε. Με την παρέμβαση τη κυρία Δαμανάκη ολοκληρώνουμε αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξή μα και η ψήφιση της, ε, των αντίστοιχων προτάσεων ψηφίσματος ε, θα γίνει αύριο στις 12 το μεσημέρι. Και περνάμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη που είναι η έκθεση της κυρίας Εντίτε Εστρέλα για την συνεργασία με τι αναπτύσσοντε χώρε όσον αφορά την πρόοδο τη χρηστή διακυβέρνηση. Συγγνώμη, για τη μείωση των ανισοτήτων στο τομέα τη υγεία. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντα ε, του γιώθει εισηγητέ ε, για τη συνεργασία και τη δουλειά που κάναμε από κοινού. Επίση, ε, του γιώθει εισηγήτρια από την Επιτροπή τη Εσωτερική Αγορά και των Δικαιωμάτων των Γυναικών, διότι όλε οι συνεισφορέ υπήρξαν ιδιαίτερα χρήσιμε. Οι ανισότητε στον τομέα τη υγεία ποικίλουν από χώρα σε χώρα από περιοχή σε περιοχή. Έχουν να κάνουν με τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες και μπορεί να επιδεινώνονται ε, λόγω φύλου ή λόγω πολιτιστικών αιτίων. Ε, αυτό σημαίνει ότι οι ανισότητες στον τομέα της υγείας έχουν ε, να κάνουν όχι μόνο με την πρόσβαση στην υγειονομική περίθυλψη, αλλά πολλές φορές και με στοιχεία και τόσο συγκεκριμένα όπω οι συνθήκε διαβίωση, η στέγαση, η μόρφωση, το επάγγελμα, το εισόδημα και ο τρόπο ζωή. Πέραν τη μερική πρόοδου που έχει επιτελεστεί υπάρχουν ακόμα μεγάλε ανισότητε στα 27 κράτη-μέλη. Για παράδειγμα, σύμφωνα με, την, με τον Eurostat το 2007, το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση παρουσιάζει διαφορά 14,2 ε, ετών μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περίπτωση των ανδρών και 8,3 έτη στην περίπτωση των γυναικών. Η υγεία και το προσδόκιμο ζωής συνδέονται επίσης και με τις κοινωνικές συνθήκες καθώς και την ένδυα, τη φτώχεια. Και επειδή η φτώχεια προκύπτει όταν υπάρχουν και άλλα ευαίσθητα στοιχεία και ομάδες όπως τα παιδιά ή οι γυρότεροι ε, ή κάποιες αναπηρίες ή το να ανήκει κανείς σε μια ομάδα που μειονεκτεί, τότε αυξάνονται και κίνδυνοι για την υγεία. Οι ανισότητες λοιπόν στον τομέα της υγείας μπορεί να ξεκινήσουν στην ε, παιδική ηλικία, να συνεχιστούν ε, στην τρίτη ηλικία και να περνούν από γενιά σε γενιά. Εξού και η σοβαρότητα του θέματος και η κατεπίγουσα ανάγκη να βρούμε μια λύση. Επιπλέον, το σημερινό γενικότερο πλαίσιο τη διεθνού κρίση έχει επιβαρύνει την κατάσταση. Όπω είναι προφανέ, αυτή η κρίση έχει σοβαρό αντίκτυπο στον τομέα τη υγεία των διαφόρων κρατών μελών και στο επίπεδο τη προσφορά αλλά και τη ζήτηση. Στο επίπεδο τη προσφορά, η κρίση μπορεί να οδηγήσει σε μείωση τη χρηματοδότηση και τη ενίσχυση του δημόσιου συστήματο υγεία, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να οδηγήσει και σε αύξηση τη προσφορά ε, υπηρεσιών υγεία. Η κρίση μας αποκάλυψε ότι η απληστία ορισμένων δεν έχει όρια και ότι αυτή η έλλειψη αξιοπρέπειας έχει συνεισφέρει στο να ε, διευρυνθεί ε, το χάσμα μεταξύ της μειονότητας των πλουσιότερων και της ε, πλειοψηφίας των φτωχότερων. Γι' αυτό η κρίση μπορεί να γίνει μια ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε τις ανισότητες μέσω μέσων τολμηρών που να προωθούν την ισότητα. Εάν τώρα δεν αντλήσουμε το δίδαγμα που οφείλουμε να αντλήσουμε και περιοριστούμε στο να αλλάξουμε ένα μικρό στοιχείο αλλά όλα να παραμένουν τα ίδια, τότε πραγματικά θα αυξήσουμε τι ανισότητε. Όμω, όπω έχουμε δει, οι κοινωνίε που δεν διαθέτουν την ισότητα είναι κοινωνίε που δεν είναι σταθερέ. Ορισμένα κράτη-μέλη έχουν συμπεριλάβει στα προγράμματά του για την ε, οικονομική ανάκαμψη ορισμένα μέτρα που σκοπό έχουν να αμβλύνουν τον αντίκτυπο τη οικονομική κρίση στον τομέα τη υγεία, επενδύοντα τι υποδομέ, βελτιώνοντα τι σηματοδοτήσει. και επαναδιοργανώνοντα το σύστημα τη υγειονομική περίθαλψη. Είναι ζωτική σημασία η αντιμετώπιση των ανισοτήτων να θεωρείται μια προτεραιότητα σε όλα τα επίπεδα τη πολιτική δράση. Για αυτού του λόγου χαιρετίζω τι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα εντωμεταξύ να πιστέψω την προσοχή σα σε ορισμένε προτάσει τη δική μου έκθεση. Πρώτα απ' όλα, ε, σε προτάσεις που στοχεύουν να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στις ανάγκες των πολιτών που βρίσκονται σε συνθήκες φτώχειας, στα, στις μειονεκτούσες ομάδες των μεταναστών και εδώ να συμπεριλάβουμε τους λαθρομετανάστες ή τις εθνικές μειονότητες, αυτούς που έχουν αναπηρίας, τους, ε, τα, τους και τα φτωχά παιδιά. Εδώ επίσης θα πρέπει να προωθήσουμε μέτρα για να αμβλυνθεί ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στον τομέα της υγείας με επενδύσεις στις υποδομές τη δημόσια υγεία. Επίση, χρειαζόμαστε συνθήκε ζωή ε, που να εξασφαλίζουν υγεία στα παιδιά και τι εγγύου. Επίση, θέλουμε να μειωθούν οι ανισότητε στον τομέα τη υγεία μέσω ε, προγραμμάτων που να επιτρέψουν να δημιουργηθεί ένα κοινό επίπεδο υγείας σε όλη την Ευρώπη. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα καλύτερο μέλλον για όλους τους συμπολίτες μας. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Ιστρέλα εννέα αγορητές. Γίνεται αυτό το οποίο συνέβη και με την προηγούμενη συζήτηση σε σχέση με την Παγκόσμια ημέρα γυναικών. Ουσιαστικά μόνο γυναίκες παρεμβαίνουν σε τέτοιες συζητήσεις και είναι σπάνια η παρουσία ενός άνδρα. Θα δώσουμε τον λόγο στην κυρία Ροϊτόβα. Κάθε μία από τις κυρίες θα έχουν ένα λεπτό για την παρέμβασή τους. Η κυρία Ροϊτόβα πρώτη. Eh, ε, Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτέ, τα τελευταία χρόνια παίξαμε πολύ σημαντικό ρόλο για να στηρίξουμε τα υγειονομικά μέτρα και την εξίσωση της κατάστασης μεταξύ χωρών μελών. Παρ' όλα αυτά, ευθελήσαμε πάντοτε να εφαρμόζεται η αρχή της επικουρικότητας. Στο 25 όμως απορρίπτω την διατύπωση. Δεν πρέπει εδώ να συμπεριλάβουμε τον έλεγχο των γεννήσεων. Όσο για το 53 και το 29, αυτά είναι αντιφατικά μεταξύ τους. Οι διαφορές στο προσδόκιμο ζωής μεταξύ χωρών της Ένωσης δεν οφείλονται εξ ολοκλήρου στην υγειονομική κατάσταση και περίθαλψη, αλλά γενικότερα στο βιωτικό επίπεδο και στην ανάπτυξη της κάθε χώρας. Και αυτό θα έπρεπε να Σας ευχαριστούμε, συνάδελφε. Η κυρία Τικάου, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η τωρινή χρηματοοικονομική κρίση έχει πλήξει και τον τομέα της υγείας. Κάποια κράτη-μέλη αποφάσισαν να κλείσουν νοσοκομεία που βρίσκονται σε μικρές πόλεις ε, ή που έχουν και μικρό αριθμό ε, ασθενών ή απομακρυσμένες περιοχές, ασθενείς από απομακρυσμένες περιοχές πρέπει να καλύψουν μεγάλες αποστάσεις ε, για να προσφύγουν σε υπηρεσίες υγείας. Υπάρχουν ανισότητες στα συστήματα υγείας που βρίσκονται στα κράτη-μέλη και μεταξύ των κρατών μελών επιπλέον η μείωση των κονδυλίων ε, για τα προγράμματα υγείας στα κράτη-μέλη προκαλούν ε, ανεπαρκείς θεραπείες. Ε, επίσης, σε σχέση με κάποιες θεραπείες, τα λυπή κονδύλια σημαίνουν ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν τη θεραπεία τους τέτοιοι πολίτες. Επίσης, αναγκάζονται να μετακινούνται από ένα κράτος μέλος σε ένα άλλο κράτος μέλος οι ιατροί για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες τους. Η κυρία Φιγκερέδο, παρακαλώ στη συνέχεια. Ευχαριστώ Πρόεδρε η σημερινή κατάσταση των πολιτικών λιτότητας, κυρίως αντικοινωνικών πολιτικών με περικοπές δημοσίων κονδυλίων ιδιαίτερα στην υγεία αυξάνουν τις ανισότητες όσον αφορά την υγεία. Όταν εξ ε, όταν λόγω των αναγκών βλέπουμε ότι αυξάνονται τα ποσοστά ε, πρόσβασης ε, στις υπηρεσίες ιδιαίτερα και για τα φάρμακα για χρόνιες παθήσεις και λόγω της μειούμενη συμμετοχή του δημοσίου και βλέπουμε και σε σχέση και με τη μεταφορά ακόμα των ασθενών σε σχέση με ζώνε που δεν υπάρχουν δημόσιε μεταφορέ, επιδεινώνονται 200 ανισότητε ανισότητες στον τομέα τη υγεία. Αυτά συμβαίνουν σε κάποια κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. ιδιαίτερα στη δική μου χώρα, την Πορτογαλία. Τα, κράτη που τα άτομα που έχουν χαμηλά εισοδήματα αντιμετωπίζουν ιδιαίτερε δυσκολίε για την πρόσβαση στι υπηρεσίε Υγεία. Γι' αυτό, κυρία Επίτροπε, κύριε και κύριοι, δεν υπάρχουν τα λόγια. Είναι αναγκαίο. Σα ευχαριστώ κυρία Φιγκερέντο, έληξε ο χρόνο σα. Τώρα θα λάβει τον χρόνο η κυρία Ζαβόσκα, παρακαλώ. Συγγνώμη, η κυρία Σίνκλερ, η κυρία Σίνκλερ θα λάβει τον λόγο, λέγει ο πρόεδρος, όχι η κυρία Ζαμπόσκα. Ε, ε, Ευχαριστώ, πρόεδρε. Η υγειονομική περίθαλψη θα πρέπει να είναι πρωταρχική με έρευνα κάθε κρατό μέλου. Διότι, όπω προτείνει και η έκθεση αυτή, χρειάζεται μια συνολική ε, ένα συνολικό σχεδιασμό για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αν, κοίταξα, αν κοιτάξετε χθε τι εφημερίδε, θα βλέπατε του Times του Λονδίνου χθε που έλεγαν για τα, τα, τα, προνόμια τα υγειονομικά των βουλευτών και την έκπτωση που έχουν κάποιε φορέ στην υγειονομική περίθαλψη. Υπήρξε 6% συνολική αύξηση του κόστου τη υγειονομική περίθαλψη μόνο πέρυσι. Εδώ μιλάμε για την ανισότητα και τις γυναίκες πολλές φορές. Ένα χαρακτηριστικό δεδομένο είναι πολύ χαρακτηριστικό. Βλέπουμε ότι... Σας ευχαριστούμε συνάδελφε. Τώρα πραγματικά θα λάβει τον λόγο η κυρία Ζαμπόσκα παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Όλοι οι άνθρωποι, κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Έχουν διαφορετικά προσόντα, δεξιότητες, τρόπο ζωής ο κάθε άνθρωπος αυτό οδηγεί τους ανθρώπους να βελτιώσουν τη ζωή τους και αυτό οδηγεί, είναι το ελαττήριο της οικονομίας. Σε σχέση με την υγεία πρέπει να λάβουμε περισσότερο υπόψη τους ανθρώπους και όχι τόσο την οικονομία διότι στις ασθένειες και στις παθήσεις είναι ίσοι οι άνθρωποι και πρέπει ισότιμα να αντιμετωπίζονται και σε σχέση και με τον όρκο του Ιπποκράτη έτσι πρέπει να αντιμετωπίζονται και όχι ως αντικείμενο κέρδους ε, το δικαίωμα για την ε, ε, έκτρωση που εμπεριέχεται στην έκθεση υποβαθμίζει αυτές τις αρχές ε, και υποχρεωτικές δυνατότητες εκτρώσεων και επιδοτούμενες κιόλας με δημόσια κονθήλια όλα αυτά δημιουργούν μια κατάσταση αφόρητη. Ευχαριστώ. Τυρίλο παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συνάδελφοι, σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθούν να υπάρχουν υγειονομικέ ανισότητε, ιδίω ό,τι αφορά την πρόσβαση στι υπηρεσίε, την περίθαλψη και του κοινωνικού παράγοντε που απαιτούν μια ολοκληρωμένη απόκριση στου υγειονομικού κινδύνου. Είναι σε πολλές περιπτώσεις ε, άδικες οι διαφορές αυτές, διότι ορισμένοι πολίτες δεν έχουν τα οικονομικά μέσα για την ε, περίθαλψη που τους αξίζει. Έτσι λοιπόν το να μειώσουμε τις ανισότητες αυτές είναι, πρώτη, είναι ζωτική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενσωματώνοντας την ισότητα σε όλες τις πολιτικές και ε, κάνοντας ισότιμη την πρόσβαση στην περίθαλψη για όλους τους πολίτες. Το Ευρωκοινοβούλιο θα παρακολουθήσει την αναθεώρηση τη οδηγία λοιπόν για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και νομίζουμε ότι αυτή είναι μια κατάλληλη ευκαιρία για να καταλήξουμε σε έναν ενισχυμένο μηχανισμό. Εκτός Τώρα θα λάβει τον λόγο ο κύριος Κέλλη, παρακαλώ. Ε, There are a number of aspects here. One... Εδώ υπάρχουν πολλές σημαντικές πτυχές. Ήθελα να σταθώ στο εξή. Ότι ο καλύτερος τρόπος να εξαλείψουμε τις ανισότητες στην οικονομική περίθαλψη είναι να κάνουμε τους ανθρώπους υγιέστερους. Βλέπω ότι πολλοί συνάδελφοι, όπως και εγώ, στηρίξαμε μια γραπτή δήλωση του Κοινοβουλίου ώστε να γίνουν μέσω του αθλητισμού και άλλων τρόπων πιο δραστήριοι άνθρωποι και πολίτες γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2020. Στην δική μου χώρα έχει δημιουργηθεί ένας συνασπισμός του ΕΛΚ και των σοσιαλιστών με όπου σκοπός της ομάδας και της πρωτοβουλίας μας είναι να συγκεντρωθούν κονδύλια για την προστασία του ασθενούς, άσχετα με τα οικονομικά του μέσα, αλλά κυρίως με βάση τις ανάγκες του. Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε κύριε Κέλλη. Τώρα θα λάβει τον λόγο η κυρία Κάρενμπαχ, παρακαλώ. Κυρία Πίτροπε, κύριε Πρόεδρε, το θέμα έχει τίτλο μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας. Και είναι φιλόδοξος στόχος. Στην σημερινή κατάσταση φοβούμε περισσότερο εμείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο παντού συνεισφέρουμε αυτές οι ανισότητες, αυτές οι διαφορές τα επόμενα χρόνια και δεκαετίες να αυξηθούν. Διότι δεν πρόκειται μόνο για οπισθοχωρήσεις όσον αφορά τον τομέα της υγείας γενικά, αλλά πρόκειται για το ποιες κοινωνικές προδιαγραφές μειώνουμε που δυσχεραίνεται η πρόσβαση, η προσπελασιμότητα στην εκπαίδευση, στην κατάτηση, εκεί όπου υπάρχουν κοινωνικές δυσκολίες ε, και τέτοια εμπόδια στην κατάτηση και παιδεία, υπάρχει φτώχεια και η φτώχεια δημιουργεί ασθένειες, ε, κάνει τους ανθρώπους να αρρωσταίνουν. Και εδώ σε σχέση με τον εθνικό προπολογισμό, τους εθνικούς προπολογισμού και τον ευρωπαϊκό προπολογισμό πρέπει να τα δούμε αυτά σε σχέση με το κόστος ε, το οποίο προκαλείται στο μέλλον. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ συνάδελφε Κάδενμπαχ. Τώρα θα λάβει τον λόγο η κυρία Αντωνέσκου, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι υγειονομικές ανισότητες είναι μεγάλη απειλή για τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξασφαλίσει ίσες δευκαιρίες, ίσα δικαιώματα και συνεκτικότητα συνοχής στις πολιτικές της. Θα έπρεπε λοιπόν αυτή η ισότητα να είναι μέρος όλων των ευρωπαϊκών πολιτικών. Θα πρέπει εδώ να συμπεριλάβουμε τέτοια στοιχεία σε όλα τα προγράμματα δράσης, σε όλες τις πολιτικές μας πρωτοβουλίες, σε όλη μας τη μελλοντική δράση, προκειμένου να μειώσουμε τις ανισότητες και να δημιουργήσουμε ψηλά πρότυπα προστασίας για τους πολίτες. Εδώ λοιπόν χρειάζεται να αναπτυχθούν δείκτες που να παρακολουθούν τις ανισότητες στον τομέα της υγείας και να υπάρχει και σύγκριση μεταξύ του από τι εθνικέ αρχέ, ώστε να αποτιμά την πρόοδο που έχει επιτελεστεί στον τομέα αυτό για να βελτιώσουμε τα υγειονομικά συστήματα. Επίση, ω μέρο των προσπαθειών μα να αντιμετωπίσουμε τι ανισότητε στην υγεία, θα πρέπει να αναπτύξουμε και στατηγικό μηχανισμό για τους εργαζομένους προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι η πρόσληψη ιατρικού προσωπικού θα είναι επαρκής. Ευχαριστούμε συνάδελφε και ολοκληρώσαμε. Ολοκληρώνουμε με την παρέμβαση του κύριου Λούχαν παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι το κάπνισμα, τα ενοπνευματόδηποτα, θα προκαλέσουν 70% των πρόωρων θανάτων, θανάτων μέχρι το 2020. Το γεγονός ότι υπάρχει συστηματική αντιστοιχία και σχέση όσον αφορά την υγεία των ατόμων και των κοινωνικών συνθήκων καταδεικνύει ότι δεν υπάρχει ισότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας οι ανισότητε στον τομέα της υγείας δεν είναι αποτέλεσμα ατομικής επιλογής. Είναι κάτι το άδικο και μπορεί να αποφευθεί αυτή η αδικία. Και σε σχέση με τις, ε, τα άρθρα που καθορίζουν ότι η υγεία είναι ένας από τις δέκα μεγαλύτερες προτεραιότητες της Ένωσης. Όταν όμως έρχεται η ώρα της υλοποίησης στρατηγικής για την Ευρώπη, της στρατηγικής του 2020, πρέπει να έχουμε διαστρωματωμένους δείκτες που θα λαμβάνουν υπόψη την διακριτική μεταχείριση σε σχέση με αυτά τα θέματα. Ευχαριστούμε συνάδελφε. Και θα ολοκληρωθεί η συζήτηση με την τοποθέτηση της Επιτρόπου της κυρίας Δαμανάκη που θα απαντήσει στις διαφορετικές αυτές παρεμβάσεις και στην κυρία εισηγήτρια. Κυρία Δαμανάκη, έχετε τον λόγο παρακαλώ. President. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Κομισιόν είναι ευγνώμων προς το Κοινοβούλιο για τη στήριξη του για τη γεφύρωση των ανισοτήτων ως προς την υγειονομική κατάσταση μεταξύ χωρών μελών. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε την εισηγήτρια κυρία Εστρέλα. Οι ανισότητες στην υγεία μεταξύ χωρών, περιφερειών, φτωχών και πλούσιων, εθνοτικών μειονοτήτων είναι κάτι που αφορά όλες τις χώρες μέλη και πολλές φορές διευρύνεται το χάσμα αυτό. Ειλικρινά θα σας έλεγα ότι μόλις τώρα βλέπουμε τις πλήρες επιπτώσεις της κρίσης στην υγεία και στις υγειονομικές υπηρεσίες. Αρχίζουμε να βλέπουμε την ανεργία που δημιουργεί η καταπολέμηση των ελλημάτων και του χρέους. Η μείωση των ανισοτήτων αυτών είναι κάτι σημαντικό και για την ευημερία των πολιτών και για την ανάκαμψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντική πρόκληση και όπως λέει και η έκθεση του Κοινοβουλίου αυτό απαιτεί συνεργασία και δράση σε συνδυασμό με πολλούς τομείς. Η έκθεσή σας κάνει σημαντικές συστάσεις για το μέλλον. Τονίζεται ότι πρέπει να υπάρξει καλύτερη πρόσβαση στις υγειονομικές υπηρεσίες και βελτίωση της ποιότητάς τους και επίσης ότι πρέπει να δοθεί προσοχή στις πιο ευάλωτες ομάδες και να χρησιμοποιηθούν νέες τεχνολογίες με τρόπο ώστε να μειωθούν και έτσι οι ανισότητες. Η Κομισιόν συμμερίζεται απόλυτα τις ε, ανησυχίες αυτές. Τονίζεται επίσης το θέμα της άνησης μεταχείρισης των φύλων και ως προς την υγεία. Προσωπικά συμφωνώ. Η Κομισιόν λοιπόν θα προωθήσει εντατικά το πρόγραμμά της για να μειωθούν οι υγειονομικές ανισότητες όπως είπαμε στη σχετική μας ανακοίνωση και σε συνεργασία και εταιρικέ σχέσεις με όλους τους ενδιαφερόμενους και κράτη-μέλη. Για να γίνουν όλα αυτά όμως πραγματικά οι χώρες μέλη αρχίζουν τώρα να εφαρμόζουν τα πρώτα τους προγράμματα με την καινούργια αυτή χρηματοδότηση που θα συμπεριλαμβάνει αξιολογήσεις τη δημιουργία περιφερειακών δικτύων και πρωτο, προώθηση πρωτοβουλειών των ενδιαφερομένων περιφερειακά. Καταρχήν ως προς την δημόσια υγεία όπως τον έλεγχο της κατανάλωσης καπνού. Η στρατική μας όμως συμπεριλαμβάνει επίσης και δεσμεύσεις σε τομείς όπως την απασχόληση και την κοινωνική πολιτική, τη γεωργία, την έρευνα και την περιφερειακή πολιτική. Προφανώς χρειάζονται περισσότερα, αλλά επίσης αυτά δεν πρόκειται να γίνουν από τη μια μέρα στην άλλη. Θα χρειαστούν χρόνια ολόκληρα για να πετύχουμε το στόχο αυτό, αλλά μπορούμε από κοινού και πρέπει να το κάνουμε ώστε να υπάρχει κάτι το απτό και να μπορέσουν όλοι οι Ευρωπαίοι να ζουν με σωστό υγειονομικό επίπεδο. Σα ευχαριστούμε κυρία Επίτροπε. Με αυτή την παρέμβαση ολοκληρώνεται η συζήτηση αυτού του θέματο. Η ψήφιση των αντίστοιχων προτάσεων ψηφίσματο θα γίνει αύριο το μεσημέρι 12.00. Και περνάμε στην ακόλουθη έκθεση.